Dear colleagues. Συνάδελφοι. Ακούσατε τα φρικτά νέα και φλιβερά ταυτόχρονα από το αεροδρόμιο των Βρυξελών. Υπήρξε μια τρομοκρατική απόπειρα, τα πράγματα εξελίσσονται και τα παρακολουθούμε. Έχουμε σοκαριστεί από αυτά που συμβαίνουν. Εκφράζουμε τη θλίψη μας και την αλληλεγγύη μας με τις, τα θύματα και τις οικογένειες τους. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στη συνεδρίασή μας αλλά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην κατάσταση και νομίζω ότι το Κοινοβούλιο στο σύνολό του θα αντιδράσει. αφού αξιολογήσει τα στοιχεία. Λοιπόν, θα σταματήσω για το συγκεκριμένο θέμα αυτό, εδώ, και θα ξεκινήσουμε με την αποδοχή των πρακτικών, τη ημερήσιας διάταξης, συγγνώμη, Α, έχουμε ένα επιπλέον σημείο. με την κατεξουσιοδότηση πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Πρέπει να εγκρίνουμε και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. 15ης, 18ης, 20ης Μαρτίου. Αύριο από τις 9.30 έχουμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Στα πλαίσια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της Ευρωζώνης. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και η Επιτροπή μας θα οργανώσουμε μια ακρόαση έτσι ώστε οι εθνικές αρχές ε, για τον ανταγωνισμό να καταστούν πιο αποτελεσματικές. Στην ιστοσελίδα μας θα δείτε την ημερήσια διάταξη. Μπορεί κανείς online να δηλώσει τη συμμετοχή του. Λοιπόν, αυτά για τις ανακοινώσεις. Περνάω στο σημείο 4. Ξεκινάμε λοιπόν την ακρόση με την Ντανιέλ Λουί της ελεγκτικής, ε, ε, του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι σημαντική η συνάντησή μας. Θα παρουσιάσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τη δεύτερη ενδιάμεση έκθεση για το SSM, όπως προβλέπεται στη Διοργανική Συμφωνία. Και εδώ καλύπτονται και οι ε, ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως ξέρετε, στην τελευταία Ολομέλεια ε, γκρίναμε την τελευταία έκθεση για την ε, Τραπεζική Ένωση η οποία εν πολλής ε, ασχολείται και με τις δραστηριότητες του SSM. Είναι λοιπόν η συγκυρία νομίζω πρόσφορη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση της κατάστασης μιας ε, λειτουργίας του μηχανισμού αυτού κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους που θα χαρακτηρίζαμε σημαντική. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι μπορώ να δώσω τώρα το λόγο στην Τανιέλ Νούι για περαιτέρω πληροφορίες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητά μέλη. Να πω ότι νιώθω κι εγώ ιδιαίτερος θλιμμένη για αυτά τα οποία συνέβησαν στο Ζάβεντεμ. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας και θα σας παρουσιάσω την ετήσια έκθεση για τις ελεγκτικές δραστηριότητες της Κεντρικής Τράπεζας για το 2015. Όταν παρουσίασα για πρώτη φορά τον μηχανισμό αυτό πέρυσι, ήταν κάτι το οποίο είχε μέλλον αλλά δεν είχε ιστορία. Στη δεύτερη έκθεση της ετήσιας αυτής παρουσίασης Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε τι έχει γίνει με την ελεγκτική αυτή εποπτική δραστηριότητα. Τώρα όχι μόνο έχουμε ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον για τον SSM, αλλά έχουμε και ένα ικανοποιητικό θα έλεγα παρελθόν. Η παρουσίασή μου σήμερα θα ασχοληθεί με τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση, κάποιες κομβικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, κάποια θετικά βήματα στην οργάνωση της ε, εποπτικής ε, λειτουργίας για επιλογές ε, από πλευράς των εθνικών διακανονιστικών πλαισίων και πριν από το τέλος θα αναφερθώ στις προτεραιότητες στον τομέα αυτό για το 2016. Ε, Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γκουαλτιέρη για μια επικοδομητική συνεργασία. Μας τροφοδοτεί με απόψεις και σημαντικά στοιχεία για το πώς βλέπει το Κοινοβούλιο ε, την κατάσταση. Να πω ποιες είναι οι γενικές εξελίξεις στον πιστοτικό τομέα. Η γενική ε, απόδοση θα έλεγα των πιστοτικών ιδρυμάτων έχει σταθεροποιηθεί μέσω της σταθεροποίησης των μακροοικονομικών συνθήκων στα πλαίσια της αποκατάστασης των προβλημάτων που δημιούργησε η κρίση. Τα πολύ χαμηλά επιτόκια δεν βοηθούν βέβαια την κερδοφορία των τραπεζών, αλλά παρόλα αυτά έχει υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αρκετά χαμηλά επίπεδα. 4,6 είναι το return on equity. Υπάρχει μια αύξηση δηλαδή σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Υπήρξαν χαμηλότερες πιστοτικές απώλειες, σταθεροποίηση επίσης των μακροοικονομικών συνθήκων. υπήρξαν στοιχεία τα οποία ενίσχυσαν γενικότερα την θέση των τραπεζών, αλλά η βιωσιμότητα αυτών των βελτιώσεων μένει ακόμα να διαπιστωθεί. Υπάρχουν αρκετά, υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία τα οποία προς το παρόν δεν μας κάνουν να είμαστε εντελώς σίγουροι υπάρχουν ε, περισσότερες διευκολύνσεις στον τομέα των πιστοτικών ικανοτήτων των τρυπεζών. Ε, η κατάσταση μπορεί να γίνει πιο δύσκολη ε, τους επόμενους μήνες. Η χαμηλή αποδοτικότητα στην ουσία πρόθεσμα θέτει σαν αμφισβήτηση ορισμένα επιχειρηματικά πρότυπα υπάρχει περιορισμένη για κάποια από τα ιδρύματα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Πάντως γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε οι τράπεζες αυτές να είναι σε θέση να αντέξουν σε κυκλικές, ε, κυκλικού τύπου εξελίξεις. Οι τράπεζες οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα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 Υπάρχει ένα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει βελτίωση του κλίματος και σε σχέση με την κήρυξη σε πτώχευση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Το 2015 οι τράπεζες σημείωσαν σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς αύξαν τα επίπεδα παροχής ε, ρευστότητας και βελτίωσαν τις διαδικασίες. Κάποια κράτη-μέλη εφαρμόζουν ε, τις απαιτούμενες διαρθρωτικές και νομικές μεταρρυθμίσεις. Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με τις ε, τράπεζες, συνεργάστηκε το 2015 για να αναπτύξει συγκεκριμένα σχέδια δράσης. Βεβαίως χρειάζεται αρκετός χρόνος για να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην εναρμόνιση των πρακτικών των τελευταίων ετών. Όπως ξέρετε το 2015 η διαδικασία, η εποπτική ονόματι ΣΡΕΠ, ΡΕΠ διεξήχθη για πρώτη φορά σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία για τις 120 μεγαλύτερους ε, τραπεζικούς ε, ομίλους ε, της Ευρωζώνης. Τα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας καθορίστηκαν από την ΕΚΤ σύμφωνα με τα προφίλ κινδύνου της κάθε τράπεζας και επιπλέον μέτρα επιβλήθηκαν όπου αυτό θεωρήθηκε αναγκαίο Επιπλέον ε, ευθυγραμμιστήκαμε με την ε, νομοθεσία και τις συστάσεις ε, διεθνών φορέων. Υπάρχει μια ολιστική αξιολόγηση όσον αφορά την εφαρμογή της αναλογικότητας. Υπάρχουν ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία μαζί με την κρίση των ειδικών. Έτσι υπάρχει μια συνέχεια και μια συνέπεια λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιαιτερότητε του κάθε θεσμικού οργάνου. Επιπλέον για πρώτη φορά επιτράπηκε, μας επιτράπηκε να υπάρχει μια συγκριτική ενιαία αξιολόγηση και άρα κάναμε ένα βήμα παραπάνω προς μια ενιαία τραπεζική αγορά. Όμως βεβαίως το θέμα είναι το πώς θα έχουμε εναρμονισμένους κανόνες λειτουργίας των τραπεζών. Όπως ξέρετε, η διακριτική ευχέρεια που υπάρχει στις υποπτικές αρχές είναι αυτή η οποία ακριβώς οδηγεί σε απόκληση των εθνικών κανόνων. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή εκεί πέρα, θα είναι αδύνατο να υποπτεύσουμε τις τράπεζες τραπεζική ένωση με τρόπο ενιαίο. Γι' αυτό ακριβώς ε, έχουμε το Συμβούλιο των Εποπτικών Αρχών και έχουμε σχεδιάσει μια εναρμονισμένη αρχή για 122 τέτοιες ε, κατευθυντήριες γραμμές στην, στην οδηγία για την κεφαλαϊκή επάρκεια υπαριθμών 4. Ε, Υπάρχει λοιπόν ένα σχετικός οδηγός Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη και τα όσα ακούστηκαν στην δημόσια διαβούλευση και εγκρίθηκαν επισήμως την προηγούμενη εβδομάδα και θα καταστούν λειτουργικά το 2016. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, αλλά οπωσδήποτε δεν είναι το τελευταίο για ίσους όρους ανταγωνισμού. Στη δεύτερη και τελευταία φάση θα εναρμονίσουμε επιπλέον 7 επιπρόσθετους τέτοιους ε, κανονισμούς για τη διακριτική ευχέρεια. Και μετά θα προχωρήσουμε στις, ε, στα λιγότερο σημαντικά τραπεζικά και πιστοτικά ιδρύματα σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ασκεί εποπτεία ολόκληρου του τραπεζικού στήματος της Ευρωζώνης και θα πρέπει να συνεχίσουμε την ε, εποπτεία αυτή. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ το τι κάνουμε στα διεθνή ρυθμιστικά φόρα για την ανάπτυξη ενός ε, διεθνούς ε, πλαισίου. συμμετείχαμε ενεργά στην Επιτροπή της Βασιλείας και εκεί πέρα συμμετέχουν οι επικεφαλής ρυθμιστικών αρχών της κάθε χώρας. Είχαμε λοιπόν τη μεταρρύθμιση της ε, Βασιλείας 3 ε, και εκπροσώπους σε διάφορες ομάδες της Επιτροπής της ε, Βασιλείας και έτσι οριστικοποιήθηκαν κάποιοι σημαντικοί φάκελοι μεταξύ των οποίων το πλαίσιο κινδύνου της αγοράς όπως επίσης και η αντιμετώπιση των θεμάτων της ολικής δυνατότητας απορρόφησης ζημιών του επιχειρησιακού κινδύνου κάποια μέτρα αύξηση της, ε, αύξησης της συγκρισιμότητας των στοιχείων των ισολογισμών των ε, τραπεζών, η αντιμετώπιση των ε, κεφαλαιακών απαιτήσεων για την τιτλοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό βεβαίως εμπλέκεστε και εσείς ως συνομοθέτης. Επίσης είδαμε το θέμα των επιτοκίων η τραπεζική εποπτεία επίσης είχε διάφορες εργασίες όσον αφορά το BCBS, την Επιτροπή της Βασιλείας, για την έκθεση των κρατών σε διάφορους κινδύνους. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στην ε, Καταρχάς έχουμε πάρει μέρος στην αντιμετώπιση του πλαισίου διαχείρισης της κρίσης επί τη βάση και του ενιαίου μηχανισμού και του BBRD. Ε, το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει με το Single Resolution Board έχει σαν στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Κεντρική Τράπεζα και τον SRM δεύτερον Προσπαθούμε σαν κεντρική τράπεζα να αξιολογήσουμε τις συγκεκριμένες τράπεζες. Μια τέτοια προσπάθεια ασχολήθηκε με εννέα τραπεζικά ιδρύματα, πέντε από αυτά δεν πέρασαν τα τεστ και η συνολική έλλειψη κεφαλαίων έφτανε το 1 δις 740 εκατομμύρια ευρώ. Ένα τμήμα από αυτά καλύφθηκε από αυξήσεις κεφαλαίου και από άλλα ε, μέτρα επιλογής στον πρώτον κύκλο των επιτόπου επιθεωρήσεων έγιναν 240 περίπου επιθεωρήσεις ε, το 2015. Ζητώ συγγνώμη. Υπάρχουν και άλλες επιθέσεις οι οποίες γίνονται και σε άλλες περιοχές ε, και γι' αυτό θα πρέπει να διακόψουμε να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. θα δούμε πώς το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει να δώσει συνέχεια. Εγώ κατανοώ ότι κάποια μέλη το χρειάζονται, αλλά αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Αυτό το οποίο ε, θέλω ε, ε, να σταματήσουμε να ζούμε. Η ζωή πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ προτείνω να υπάρξει μια προσωρινή διακοπή για να αξιολογηθούν τα γεγονότα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με τον πρόεδρο και ε, τους ε, ε, κοσμήτορες. Μπορεί να τίθενται θέματα ασφαλείας και θα σας ενημερώσω για το πώς θα συνεχίσουμε. Λοιπόν 10 λεπτά διακοπή και μετά θα επανέλθω. Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, είχα κάποιες συνεννοήσεις ε, με τους αρμόδιους εδώ του Κοινοβουλίου που παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Το κτίριο είναι ασφαλές. Και περιμένουμε κάποιο μήνυμα. Ε, μπορεί να είναι δύσκολο βεβαίως, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε την συνεδρίασή μας για να στείλουμε το μήνυμα που έλεγε η Σιλβή. Εγώ θα σας προτείνω να συνεχιστεί η συνεδρίαση και όταν λάβουμε οδηγία θα κινηθούμε αναλόγως. Τον λόγο έχει λοιπόν η ομιλήτρια. Τελείωνα. Με τις προσπάθειες που κάνουμε με την Επιτροπή των Βρυξελών, τον Brussels Committee μάλλον, και τα θέματα της, ε, του δημοσίου χρέους. Υπάρχουν και άλλα προγράμματα με τα οποία ασχοληθήκαμε το 2015 στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τον SRM Όπως είπα κάναμε πάνω από 240 επιτόπιους ελέγχους τον προηγούμενο χρόνο. Έχουμε και μια κεντρική ομάδα ελέγχου, εποπτείας, η οποία ασχολείται με την ομοιογενή εφαρμογή του συστήματος που έχει επιλεγεί. Χρησιμοποιείται ένα εσωτερικό πρότυπο μοντέλο σε κάθε χώρα για τον υπολογισμό των αναγκών σε κεφάλαια των τραπεζών. Στόχος είναι να υπάρξει εφαρμογή των προτύπων αυτών με ενιαίο τρόπο. Οι προτεραιότητες τώρα για το 2016 είναι η αξιολόγηση των κινδύνων σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές γίνεται η αναζήτηση αυτών των προτεραιοτήτων όπως και οι αναλύσεις ε, οι μικρό και μακροπροληπτικές. Ανάμεσα στους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε είναι τα επιχειρηματικά πρότυπα για την αποδοτικότητα και υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι, η σημασία των οποίων εξαρτάται από τις εθνικές αρχές. κίνδυνοι ε, διακυβέρνησης, κίνδυνοι σε σχέση με το δημόσιο χρέος, ε, ευπαθείς μορφές έκθεσης σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες. Θέλουμε γενικά να διασφαλίσουμε οι τράπεζες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά με ενιαίο τρόπο και αυτό θα χαρακτηρίζει την προσπάθειά μας για το 2016. καταλληλότητα των, της κεφαλαιοποίησης της κάθε τράπεζας, όπως επίσης και διασφάλιση της ρευστότητας σε σχέση με τις λειτουργίες της κάθε τράπεζας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ε, υπάρχει πλήρης εφαρμογή όλων αυτών των στόχων για πάνω από ένα χρόνο και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί η κατάσταση. Κλείνοντας θα έλεγα ότι ο SSM δεν είναι μόνο ένας αυστηρός επόπτης εμείς θέλουμε να συνεισφέρουμε στην ακαιρεότητα της ενιαίας αγοράς, διασφαλίζοντας ότι οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους και να τους χρησιμοποιήσουν για την ανάπτυξη. Εφόσον οι κανόνες αναχώρα διαφέρουν, αυτό είναι κάτι που δημιουργεί θέματα. Υπάρχουν βέβαια οι επιλογές οι, σε εισαγωγικά εθνικές, υπάρχουν δηλαδή οι δυνατότητες διαφοροποίησης, αλλά παρόλα αυτά αυτές οι εξαιρέσεις θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ε, δεν έχουμε πάρα πολλά περιθώρια σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέμβασης και η έκκληση την οποία απευθύνεται και εσείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ετήσια έκθεσή σας για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για περαιτέρω εναρμόνιση μας βρίσκει σύμφωνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για το πρώτο έτος αυτό δραστηριότητας και πρέπει να πω, όπως, λέτε, όπως λέμε και στην έκθεση, για τον ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, περνάμε σε ερωτήσεις. Ο Μπορκαρτ δεν εδώ. Λοιπόν, έχετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Αλλιώ περνάμε στον επόμενο μιλητή. Παύλο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και σας ε, κύρια Νουή για αυτά που μας είπατε σε μια πολύ δύσκολη μέρα στις Βρυξέλλες. Την προηγούμενη φορά που είχατε έρθει εδώ πέρα σας ρώτησα για την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ιρλανδίας για αυστηρότερους ε, μακροπροληπτικούς ε, κανόνες. Αυτή τη στιγμή βεβαίως είναι δραματική η κατάσταση στον τομέα της στέγης, ε, αυξάνονται τα νίκια, δεν υπάρχει επαρκής στέγη. Το θέμα λοιπόν είναι αν πρέπει να έχει κάποια ευελιξία η κεντρική τράπεζα, π.χ. να μπορεί να σφίγγει λίγο τα λουριά ή αντιστρόφως να χαλαρώνει αναλόγως συνθήκες. Δηλαδή πως θα έπρεπε να παίζει έναν αντικυκλικό ρόλο όπως γίνεται και με άλλους τομείς πολιτικής όπως η δημοσιονομική. Η δεύτερη μου ερώτηση είναι αν πιστεύετε πως ε, η στέγη θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως ένας δείκτης μακροπροληπτικής ε, πολιτικής. Ε, τέτοιοι δείκτες, παραδείγματος χάρη για το σφίξιμο θα έλεγα των λουριών στην πίστη θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια προσαρμογή της ε, πολιτικής των κεντρικών τραπεζών. Και τέλος, ποιοι είναι οι κίνδυνοι για τον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα εάν γίνει Brexit. Υπάρχει ο κίνδυνος να πάνε κάποια γραφεία, τα front office σε άλλες χώρες, εάν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι εάν ένα τέτοιο πιστωτικό ίδρυμα αντιμετωπίσει ζήτημα φερεγγιότητας. Ποιος θα φταίει σε αυτή την περίπτωση, το κράτος μέλος ή ο SSM και ο οργανισμός σας ο Μηχανισμός Σταθερότητας έχει κάνει μια αξιολόγηση των ε, δυνητικών κινδύνων του Brexit. Ευχαριστώ. Regarding, ε, Όσον αφορά τα μέτρα της Ιρλανδική ε, Ιρλανδικής Κεντρικής Τράπεζας τα μακροπροληπτικά Νομίζω πως είναι πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε τους πιθανούς κινδύνους όπως τα εργαστικά δάνεια ή την κρίση των ακινήτων είναι απόφαση των εθνικών εποπτικών αρχών την οποία εγώ σέβομαι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να συμπληρώσει αυτά τα μέτρα και αν θεωρούσε ότι απαιτείται κάτι τέτοιο ε, και δεν ε, γίνεται να αναλάβει μια πρωτοβουλία αλλά αυτό βεβαίως επαφίεται στις ε, εθνικές εποπτικές αρχές τις κεντρικές τράπεζες κάτι το οποίο Βεβαίω είναι σωστό γιατί υπάρχουν 19 διαφορετικοί τρόποι παροχής στεγαστικών δανείων όσον αφορά τις ε, στεγαστικές ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό ήταν ε, το πρώτο το οποίο ζήτησα από τους συναδέλφους όταν αναλάβαμε. Δηλαδή μια ταυτότητα θα έλεγα για τη στεγαστική πίστη στην ε, κάθε χώρα για να δούμε τα χαρακτηριστικά της και θα δημοσιεύσουμε μάλιστα κάτι για τα διαφορετικά είδη στεγαστικών δανείων στην Ευρωζώνη σύντομα. Ίσως και εντός εβδομάδος. Τώρα, αν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση στην στέγη για τη μακροπροληπτική πολιτική. Οπωσδήποτε, γιατί η υπερβολική προσφορά, η έλλειψη προσφοράς είναι κριτήρια τα οποία επηρεάζουν το επίπεδο των τιμών και την κατάσταση των αγορών. Οπότε λαμβάνονται υπόψη. Τώρα εγώ δεν θα απαντήσω για το εάν πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, για την νομισματική πολιτική γιατί δεν ξέρω εγώ από αυτά. Δεν ήμουν ποτέ υπεύθυνη για την νομισματική πολιτική. Ε, λειτουργούμε, ξέρετε, υπό έναν αυστήρο διαχωρισμό μεταξύ του κλάδου νομισματικής πολιτικής ε, και του εποπτικού κλάδου. Για τον Brexit τώρα δεν θα κάνω κάποια πρόβλεψη για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ούτε να υπολογίσω τις ε, δυνητικές συνέπειες. Αλλά η ερώτησή σας είναι διαφορετική γιατί αφορά την κατάσταση των ε, τραπεζών που θα μπορούσαν να πάνε στην υπηρετική Ευρώπη. Α, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα σχολιάσω μια αποθετική κατάσταση αλλά Αυτά τα έχει ρυθμίσει ούτω ή άλλω ε, ο ρυθμιστής. Ίσως έχουμε τράπεζες που είναι συστημικές ε, και ίσως απαιτήσουν περισσότερους πόρους. Και... Επίσης βλέπω και κάποια πλέον εκτήματα θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στην υπηρετική Ευρώπη. Αλλά και πάλι δεν θα σχολιάσω υποθετικές ε, καταστάσεις. Ευχαριστώ Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ. Αυτά που συμβαίνουν ε, σήμερα δεν μας επέτρεψαν να ακούσουμε με προσοχή την ε, αρχική σας παρέμβαση. Λόγω των περιστατικών λοιπόν ε, δεν δώσαμε την απαραίτητη προσοχή. Θα ήθελα λοιπόν να επανέρθετε ε, στα στοιχεία αυτά που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε τη μετάβαση από την προηγούμενη νοοτροπία του τραπεζικού συστήματος στην Ευρώπη προς μια νέα, με τη νέα με τις νέες νομοθετικές διατάξεις που θεσπίστηκαν και εφαρμόστηκαν με τη συμβολή του Κοινοβουλίου. Ε, ιδρύθηκαν νέες οντότητες. Για το θέμα που με ενδιαφέρει υπάρχει ο νέος υπεπόπτης. Υπάρχουν λοιπόν δυσκολίες σε αυτή την μετάβαση και θα ήθελα να συζητήσετε για τις ανισορροπίες που προκύπτουν ε, λόγω της αδυναμίας προσαρμογής στη νέα κατάσταση ε, λαμβάνονται δεόντως υπόψη από τον νεοπεπτοϊκό μηχανισμό. Αναφερθήκα σε διάφορα στοιχεία, αλλά συγκεκριμένα με ενδιαφέρει οι επιπτώσεις της οικονομικής παρατεταμένης ε, οικονομικής ύφεσης και του στασιμού πληθωρισμού ε, για την ε, κερδοφορία των ε, τραπεζών, την αποδοτικότητα των τραπεζών σε συνδυασμό με τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και ταυτόχρονα υπάρχουν οι απαιτήσει αύξηση τη κεφαλαϊκή επάρκεια, τη διαφάνεια και όλα αυτά ε, συνδυάζονται με τι νέε διατάξει τη Τραπεζικής Ένωσης. Όλα αυτά σε κάποιε αγορέ δημιουργούν την αίσθηση τη αστάθειας, της έλλειψης εμπιστοσύνη στο μέλλον και νομίζω ότι θα πρέπει να δυσκολιάσετε διότι δεν απορρέει, κατά τη γνώμη μου, από την Τραπεζική Ένωση αλλά από τι δυσκολίε της μεταβατικής αυτής περίοδου. Θα μπορούσατε λοιπόν ε, να μας πείτε σε ποιο βαθμό ε, υπάρχει αυτή η συνειδητοποίηση σε επίπεδο ημίου οπτικού μηχανισμού των μεταβατικών δυσκολιών δηλαδή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ, είναι δύσκολη αυτή η μεταβατική περίοδος. Αυτό εξηγεί και τις αναταράξεις των αγορών ε, στις αρχές του χρόνου. Ο παλιός χρόνος, ε, με παλιά εποχή του bailout και η νέα εποχή του bail-in. Οι επενδυτές ε, δεν συνειδητοποιούν πλήρως άμεσα τη νέα κατάσταση και τις επιπτώσεις που αυτή έχει για αυτούς. Φυσικά, έχουμε πλήρη επίγνωση της κατάστασης Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε ευελιξία για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε. Χρειαζόμαστε χρόνο για να ληφθούν όλα αυτά τα νέα δεδομένα υπόψη. Παραδείγματο χάρη, αναφερθήκατε στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μα χρειάζεται χρόνο για να επιδιορθώσουμε την κατάσταση για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις πτυχές του προβλήματος. Χάρη όμως στη συνολική ε, ε, αναθεώρηση ε, με τον κοινό ορισμό από τον Παϊμπά εντοπίσαμε όλα τα κόκκινα δάνεια και έχουμε επαρκή αποθεματικά για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι έχουμε γερά θεμέλια ούτω ώστε με τον πλέον πρόσφορο τρόπο να αντεπεξέλθουμε στα προβλήματα. Νομίζω πως ε, αντιμετωπίζουμε <clears throat> όλα αυτά τα ζητήματα λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που προκύπτουν Είναι πλήρω εφικτό πάντω ότι έχουμε ασφαλεί και υγιεί τράπεζε σε όλη την Ευρώπη. Θα το πετύχουμε. Χάρη στι προσπάθειε των ε, εθνικών εποπτικών αρχών ε, που μα προσφέρουν ε, την εμπειρία, τι γνώσει, δεξιότητε που έχουν. Έχουμε και το πλαίσιο του SSM, του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Και έχουμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας για να ληφθούν ε, οι κατάλληλες αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι προς το παρόν έχετε λάβει όλη την πρώτη ανακοίνωση από το DigiSafe που λέει ότι αυξάνεται το επίπεδο ασφαλείας στο πορτοκαλί για τα κτίρια Μα ζητούν να παραμείνουμε μέσα στο κτίριο και θα μας ενημερώσουν. Ο Μπέντ Λούκα. Θέλω να μιλήσω γερμανικά. Το ερώτημά μου αναφέρεται στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αναφέρατε. Σωστά είπατε πως έχουν διαφορετικές αιτίες μεταξύ των οποίων την γενική οικονομική συγκυρία αλλά και διαρθρωτικές αιτίες όσον αφορά τους νόμους χρεοκοπίας παραδείγματος χάρη ή άλλα μέτρα διαρθρωτικά. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω το εξής. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε πως ε, μπορεί να θεωρηθεί ως ε, μία αιτία ή γενικότερη οικονομική συγκυρία. Και θα ήθελα να δούμε ακριβώς τις εξελίξεις αυτές σε σύγκριση με τις ίπα όπου το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων μέχρι το 2010 ήταν σταθερό. Από το 2010 όμως έχει τελείως διαφορετική εξέλιξη με σαφ σαφή μείωση στη ΣΥΠΑ και σαφή άνοδο στην Ευρωζώνη. Οπότε το ερώτημά μου είναι οφείλεται στις διαφορετικές μακροοικονομικές εξελίξεις που ήταν κάπως καλύτερες στη ΣΥΠΑ από την Ευρωζώνη ή θα λέγατε πως οι διαφορετικές μακροοικονομικές εξελίξεις δεν ήταν τόσο ισχυρές ε, για να επηρεάσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το δεύτερο ερώτημα αφορά αυτό το οποίο είπατε για τους νόμους περί χρεοκοπίας και ως έναν διαρθρωτικό παράγοντα. Δεν έχω καταλάβει πώς το εννοείτε. Υποθέτω πως παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια εφόσον δεν τα έχει διαγράψει κάποια τράπεζα και δεν έχει παρετηθεί από την απέτηση. Βεβαίως μια τράπεζα όπως είπαμε μπορεί να τα διαγράψει και να αποδεχτεί την οικονομική πραγματικότητα ακόμα και αν νομικά εξακολουθεί να έχει τις απαιτήσει. Οπότε μετά τίθε το ερώτημα μήπως θα έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια πολιτική διαγραφής των μη εξυπηρετούμενων δανείων από του ισολογισμού των τραπεζών. Και μετά τίθεται το ερώτημα σε εσά στην εποπτική αρχή, μήπως ε, το θεωρείτε αυτό δουλειά σας ε, δηλαδή να προχωρήσουμε σε μια πιο έντονη διαγραφή από του ισολογισμού των ε, δανείων αυτών. Και τι θα συνέβαινε σε αυτή την περίπτωση. well, οι NPL είναι εξυπηρετούμενα δάνεια ε, ε, ανεξαρτάται αν ε, μιλάμε για εταιρείε, ε, για μικρομεσαίες, για ιδιώτες, εξαρτάται από το νομικό περιβάλλον δεν είναι μόνο οι οικονομικές ε, οι παράμετροι που επηρεάζουν ε, την κατάσταση. Υπάρχουν και άλλες. Ε. Ως επιτοπλίστων βέβαια είναι οικονομικό ζήτημα, αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλες τις λύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. το ειδικό πλαίσιο εγγυήσεων που ε, ε, θέσπισε η Ιταλία παραδείγματο χάρη η πώληση των στοιχείων ενεργητικού σε ειδικού επενδυτές ε, που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση ή ξεκαθάρισμα του ισολογισμού των τραπεζών, ε, ποια δάνεια μπορούν να τα αναδιαρθρώσουν και ποια όχι. Επειδή είναι μη εξυπηρετούμενα και θα πρέπει να καταλογιστούν ως ε, ζημιά. Οι ζημιές ή αδυναμία ανάκτησης εγγυήσεων, ε, παραδείγματος χάρη, γιατί πριν από λίγο καιρό αυτό συνέβη σε κάποια κράτη. Δεν μπορούσαν νομικώς να ε, επανακτήσουν τις εγγύησεις. δεν, ε, ορισμένες φορέ δεν είναι ότι δεν χρησιμοποιούν τα ειδικά μέσα που έχουν, Απλώς δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες. Όμως τώρα αυτό βελτιώνεται. Το προσωπικό είναι σε πολύ καλύτερη θέση σήμερα για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Ορισμένες φορές ε, δεν ε, είναι αρκετά ποιοτικά τα μέσα που έχουν ε, στη διάθεσή τους. Τώρα δεν ξέρουμε καθόλου σίγουρη αν ένα ενίο εργαλείο, μια ενιαία λύση μπορεί να δώσει απάντηση σε διαφορετικές ε, περιπτώσεις, ε, για διαφορετικούς ε, δικαιούχους, για διαφορετικά, διαφορετικές καταστάσεις στα κράτη-μέλη. νομίζω ότι Α, γιατί η δημοσίευση των πληροφοριών ε, δεν γίνεται να έχουμε υγιείς και ασφαλείς τράπεζες αν δεν υπάρχει κοινοποίηση στοιχείων. Γιατί ο στόχος είναι να αποπληρώνεται το δάνειο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και ε, όλες τις καλές συμβουλές ε, τις θεωρούμε πραγματικά ευπρόσδεκτες στην εργασία με το δούνο του. εμπνεόμαστε από τις ε, υποπτικές ε, παραδόσεις, υποπτικές πρακτικές των κρατών μελών με, τα οποία συνεργαζόμαστε. Ευχαριστούμε Σιλβί Γκουλά. Ευχαριστώ που μας επιτρέψατε να συνεχίσουμε. Ε, είχε νόημα η διακοπή, αλλά για μια ακόμη φορά πρέπει να πω ότι εμείς μπαίνουμε σε μια περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας πρέπει να, να υπερασπίσουμε αυτά στα οποία πιστεύουμε. Ίσως, ε, Ντανιέλ, να έχεις ε, δυσκολία να επιστρέψει στη Φραγκφούρτη, οπότε θα εκμεταλλευτούμε την παρουσία σου εδώ. Ε, θα ήθελα να πω με πραγματιστικό τρόπο, τι πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε στη σχέση σας με την EBA. Ίσως υπάρχουν και κάποιες σκέψεις για το τι θα γίνει με τις επενδυτικές τράπεζες και με τις ασφαλιστικές εταιρείες. Και δεύτερον, θα ήθελα να μου πείτε αν συμμερίζεστε αυτό το οποίο νιώθουμε το τελευταίο καιρό κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τη Μεγάλη Βρετανία, ότι η ζώνη ευρώ δημιουργεί θέματα στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς γιατί οδηγεί τις χώρες που δεν ανήκουν στη ζώνη ευρώ σε μια μειοψηφική αν θέλετε κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι η ζώνη ευρώ αντίθετα ενιοποιεί τις θέσεις των χωρών και μήπως τελικά αυτοί οι οποίοι μένουν εκτός της ζώνης ευρώ φύγουν την ποιότητα της ενιαίας αγοράς και φύγουν και υπονομεύουν την ποιότητα των κανόνων μας και στον πιστοτικό τομέα που θα ήθελα να είναι όσο πιο ενιαίοι γίνονται οι κανόνες αυτοί. θα πρέπει να απαντήσω στα αγγλικά για να με καταλάβετε. Λε κυρία Νουί; Σχετικά με την αναθεώρηση της εποπτείας του SSM. Αναφερθήκατε επίσης και στην EBA και έχουμε πολύ καλές σχέσεις με αυτό το όργανο και με την Ιούπα όπως λέμε στα γαλλικά είμαι από τους παλιούς σε αυτές τις επαφές έχουμε συζητήσει μαζί τους επανειλημμένα στο παρελθόν δεν υπάρχει εδώ σύγκρουση συμφερόντων σε ό,τι με αφορά αλλά για να μπορέσουμε να ακουστούμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση Είναι περίεργο το ότι οι πρόεδροι της ΦΕΜΠΑ και της ΙΟΠΑ δεν έχουν δικαιώματα ψήφου. Κάποιον βλέπω εδώ, λέει ο πρόεδρος, από τα δύο αυτά όργανα. δεν έχουμε κι εμείς δικαίωμα ψήφου. Στην EBA είμαστε παρατηρητές, όλα αυτά έχουμε εξαιρετικές σχέσεις. Υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ακόμα και αν όπως είπα δεν έχουμε δικαιώματα ψήφου. αυτό το οποίο γίνεται ότι κάθε μικρή έστω λεπτομερής απόφαση πρέπει να ληφθεί σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου. Πρέπει να συντάσσουμε συνεχώς σημειώματα, μικρά κείμενα. Δεν είναι ακριβώς αυτή η εποπτική δραστηριότητα. Έχουμε και ζώνες όπου δεν είναι προφανές το τι πρέπει να κάνει και ποιος πρέπει να το κάνει. Υπάρχει ακόμα μια σύγχυση. Υπάρχουν τομείς που είναι ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες, οι εξουσίες σε εισαγωγικά οι αρμοδιότητες του SSM είναι σαφείς και σε σχέση με τον κανονισμό που ε, θα φέρει την θέση σε εφαρμογή των ε, αποφάσεων Βασιλεία 3 αλλά πάντως υπάρχει συνολικά ουσιαστικά ένα μεγάλο δίκτυο μέσα στο οποίο ακούγονται και διαφορετικές απόψεις, σαν παράδειγμα με κάποιους εθνικούς επόπτες για το τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τι πρέπει να κάνει το SSM, τι πρέπει να κάνουν οι εθνικοί επόπτες και γι' αυτό Ε, πολλές φορές μέσω των οδηγιών που είμαστε υποχρεωμένοι να δίδουμε προς τους ε, εθνικούς επόπτες ε, στην ουσία αυξάνουμε την εργασία την οποία κάνουμε και θα μπορούσαμε ίσως να το κάνουμε και σε κεντρικό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο να βρούμε τρόπους έτσι ώστε ο τρόπος που λειτουργούμε να γίνει πιο αποτελεσματικός και εύκολος. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συμφωνήσω με την τελευταία σας παρατήρηση, ίσως να είμαι λίγο προκατηλημένη, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό η προσπάθεια η οποία γίνεται στην Ευρωζώνη να, να υπογραμμιστεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα οι διαδικασίες ε, ε, εναρμόνισης και μέσω της μεθόδου των national options των εθνικών επιλογών Όλη η προσπάθεια την οποία κάνουμε λοιπόν έχει σαν στόχο οι τράπεζες, όλες οι τράπεζες να είναι ασφαλέστερες, να είναι υγιέστερες και να συνεισφέρουν στην εσωτερική αγορά για το σύνολο της Ευρώπης. όπως είπα, ίσως, ίσως είμαι λίγο προκατηλημένη, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι το θαυμάσιο η Ευρωζώνη και θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους και οι χώρες που είναι εκτός. Δεμάζει. Yeah, uh, allows... Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα και εγώ να μιλήσω γερμανικά. Συλληπιτήρια και από μένα Δεν είμαστε ανέστητα μοσχάρια βεβαίω. απλά συνεχίζουμε να δουλεύουμε γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Λοιπόν, υπήρχε μία συνεννόηση με τα κρατήρια του Αμβούργου και του Σλεσβιχ Χόλσταϊν για κάποια μη εξυπηρετούμενα δάνεια και θα πρέπει να αναλάβουν τα κρατήδια ε, γύρω στα 3 δισεκατομμύρια και είχα Χασάς να αναλάβει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια από τις υποχρεώσεις αυτές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει μια μείωση από την τιμή αγοράς γύρω στα 40% έχουμε αυτή την εγγύηση η οποία όμως ήδη έχει γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση και βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, όλα αυτά έχουν πάρα πολύ χαμηλή τιμή αγοράς ε, και έτσι θα μπορούσε να μην ε, ισχύει πια η εγγύηση. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση. Και... Και ποια είναι η άποψή σας ε, για την δυνατότητα της τράπεζας αυτής της Χάντζα χωρί για να μπορέσει να επιβιώσει. Και βεβαίως ε, βλέπετε κάποια ανάγκη διόρθωσης ε, Επίσης για τα ομόλογα τα κόκος βλέπουμε τις εξελίξεις ε, και στην Ιταλία όπου κινδυνεύουν οι οικονομίες των ανθρώπων. Βλέπετε κάποιο πρόβλημα στην εποπτεία των τραπεζών και τι συμπεράσματα βγάζετε για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. γιατί υπάρχει βεβαίως ε, και το ζήτημα αυτό των τραπεζών του Big to Fail. Ο πρόεδρος. Κοιτάξτε, ε, δύο λεπτά τώρα η ερώτηση πρέπει λίγο να περιοριστείτε κάπως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εάν κατάλαβα καλά, το πρώτο τμήμα της ε, ερώτησής σας Μιλάτε για μια γερμανική τράπεζα η οποία συζητά κάποια σχέδια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάποιες εγγυήσεις που ήταν στο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω συγκεκριμένα πιστοτικά ιδρύματα. Μάλιστα χτες όταν έφυγα από τη Φραγκφούρτη ε, οι διαδικασίες ε, συνεχίζονταν οπότε δεν ε, μπορώ να σε ενημερώσω για τις πιο τελευταίες εξελίξεις. Αλλά είμαι σίγουρη ότι η τράπεζα σύντομα θα ενημερώσει τις αγορές. Γιατί κάτι είδα με το, στο Blackberry ερχόμενοι στις Βρυξέλλες. για τα stress test τα οποία κάνουμε να μιλάτε για αυτή την συνολική αξιολόγηση εμείς θεωρούμε ότι κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά γίνεται για όλες τις ε, τράπεζες ε, που είχαν κίνδυνο δεν ανακαλύψαμε μέχρι στιγμής κάποια προβλήματα στην αξιολόγηση την συνολική. Ούτε κάναμε το σενάριο για τις ανερχόμενες ε, οικονομίες. Α, ναι, ναι, ναι, αυτό μου ξέφυγε. Κοιτάξτε. Το σενάριο αυτό το δυσμενές το ψηφίζουν τα μέλη της EBA ε, όπου εμείς δεν έχουμε ψήφο και μετά το εγκρίνει η Εκτελεστική Επιτροπή του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. Αυτά δεν τα εγκρίνουμε εμείς, αλλά όσοι ασχολούνται με την οικονομική κατάσταση. Οπότε δεν τα κάνουμε εμείς αυτά. Όσον αφορά τα κόκκος, τα οποία πολλούνται σε πελάτες λιανικής. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι η προστασία των καταναλωτών. Ήμουν αρμόδια για αυτό το θέμα. Δεν είμαι πια. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε αλλά πράγματι τα μέσα αυτά τα αγοράζουν οι πελάτες γνωρίζοντας τι είναι. Κοιτάξτε τώρα για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα γιατί οι τράπεζες παίζουν μεγάλο ρόλο στην Ευρώπη, στη χρηματοδότηση της οικονομίας. 70% της χρηματοδότησης παρέχεται από τις τράπεζες και 30% από τις αγορές στις ΕΠΑ ΕΕ είναι το αντίστροφο. Οπότε χρειάζεται μια διάσταση δημιουργίας αγοράς ε, για να βοηθήσουμε τις εταιρείες να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Αυτό σημαίνει πως ε, πιθανότατα θα πρέπει να συνεχίσει αυτή η δημιουργία αγοράς ε, με τις ε, λειτουργίες λιανικής ε, τραπεζικής και να μην ε, πάει με το κομμάτι, με το κομμάτι επενδυτικών τραπεζών αν υπάρξει διαχωρισμός όπως είδαμε με κάποιες γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Υπήρχε όπως είπαμε κάποια δημιουργία αγοράς γιατί όπως σας είπα δεν είχε ακόμα ψηφιστεί πλήρως ο διαχωρισμός αλλά προφανώς ε, η διαφορά μεταξύ της φετινής αναταραχής και των προηγούμενων ετών είναι ότι η αναταραχή αυτή αφορούσε λιγότερους δημιουργούς αγοράς. Ε, και ήταν πραγματικά κτηνώδεις δύσκολες αγορές Στην παράγραφο 11 της έκθεσής μας ε, λέει γιατί τα ε, διδάγματα που αντλήσαμε από τις ε, αναθεωρήσεις Πότε θεωρούμε ότι είναι υγιής το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πότε χρειάζεται παρέμβαση Και έχουμε και την ε, κύρια μεθοδολογία για τις εκθέσεις ε, των τρίτων χαρών επί τη, με βάση της αξιολόγησης. Ξέρουμε ότι έχετε ρόλο και στην ABA για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Yeah, it's, uh... Ευχαριστώ. είναι φοβερή σύγχυση και δεν μπορώ κιόλας να, να πολυμιλήσω με αυτά που συμβαίνουν. Τέλος πάντων, σε σχέση με αυτά που είπε ο Φάμπιο, δεν έχει εντολή προστασίας ο SSM, αλλά επειδή δεν έχουμε προστασία για τους επενδυτές και για τους καταναλωτές, αυτό μπορεί να έχει επιπτώσει επί της οικονομικής σταθερότητας και της δέουσας επιμελητίας. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω αν ε, κάνετε κάτι γι' αυτό και αν έχετε γι' αυτό εντολή. Δεύτερον, στην ετήσια έκθεση και η παρόδο να σας συγχαρώ για αυτή την πρώτη έκθεση. Στην σελίδα 32 λέτε ότι κατά 30 μονάδες βάση αυξήσατε τις απαιτήσει του πυλώνα 2 για την περίοδο 2015-2016. Δεν είναι προκυκλικό όμως αυτό, έτσι που έχουν τα πράγματα στην Ευρωζώνη και γι' αυτό θα ήθελα να καταλάβω ακριβώς πώς ε, από αυτή την άποψη συνυπολογίζεται τις διαφορετικές καταστάσεις ε, που ισχύουν στις αγορές. Ε, η Bundesbank, παραδείγματος χάρη, στην έκθεση οικονομικής σταθερότητας τόνισε ότι 30% όλων των, όλης της καταναλωτικής πίστης για τη στέγη δίνονται σε πάρα πολύ χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με την ε, αξία του ακινήτου. Επίσης από ένα γράμμα ε, ομάδας ειδικής πίεσης έμαθα ότι κάνετε ήδη σπλήτες στις απαιτήσει του δεύτερου πυλώνα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς το κάνετε αυτό. Ποια κομμάτια του ε, δεύτερου πυλώνα είναι πολύ υποχρεωτικά για το σημείο ενεργοποίηση του MDA και ποια όχι. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο δεύτερος πυλώνας έχει ένα δεσμευτικό και ένα μη δεσμευτικό κομμάτι και σε τι βασίζεστε για να κάνετε αυτό το διαχωρισμό, αυτό το split. Ευχαριστώ για τι ερωτήσει σα, για τον πυλώνα 2 και την προκυκλικότητα ή όχι των μέτρων. Κατά μέσο όρο για τις απαιτήσει του δεύτερου πυλώνα αυξήσαμε κατά 30 μονάδες βάσης φέτος τις απαιτήσει. Πρέπει να προσθέσω σε αυτό πως η δρυπτική πλειοψηφία των τραπεζών που είδαν αυτές τις αυξήσεις στο δεύτερο πυλώνα το είχαν αυτό το κεφάλαιο ήδη, οπότε δεν χρειαζόντουσαν επιπρόσθετες κεφαλαιοκικές ε, απαιτήσει. Επίσης υπήρχαν διάφορες χώρες όπου οι τράπεζες είχαν πολύ καλή κεφαλαιοποίηση και οι απαιτήσει ε, του δεύτερου πυλώνα ήταν κάπου μεταξύ των απαιτήσεων χωρίς ε, να ασχοληθούμε πολύ αν είναι 8,5 ή 9,5. Ήταν πολύ πάνω από το 10% οι τράπεζες. Για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Για τις 30 ε, μονάδες βάσης πρέπει να ξέρετε ότι έγινε κυρίως για τις τράπεζες ε, που ε, δεκάρα δεν δίνανε για τις απαιτήσει του δεύτερου πυλώνα γιατί ήταν πολύ παραπάνω αυτά που είχαν ήδη. Γιατί θέλαν στους ίσους όρους ανταγωνισμού και είχαν ήδη ξεπεράσει τα απαιτήσει, ήταν στο 9,5 ή στο 10. Τεχνική διόρθωση λοιπόν με μηδενικές επιπτώσεις. Λιγότερες από 10 ήταν οι τράπεζες ε, που δεν είχαν τις απαιτούμενες, ε, την απαιτούμενη κεφαλαιοποίηση όταν πήραμε εμείς αποφάσεις και οι περισσότεροι είχαν την κάλυψη για αυτές τις επιπρόσθετες απαιτήσει του δεύτερου πυλώνα. Δεν νομίζω λοιπόν πώς δημιουργήθηκε προκυκλικό ζήτημα. Δε, συγγνώμη, δεν... δε σημείωσα καλά τι είπατε για τη Γερμανία. Α, ναι, ναι, για τα στεγαστικά λέτε. Τα στεγαστικά, ναι. Είναι ασυνήθιστο αυτό που συμβαίνει. στο φόρουμ για τη μακροληπτική εποπτεία, όταν συζητάμε για τα μέτρα, το συζητάμε και αυτό φυσικά, το εξετάζουμε. Τα ενυπόθηκα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι των συζητήσεών μας πάντοτε, οπότε δεν έχει ληφθεί κάποια δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τελικά οι εθνικές, οι εθνικοί επόπτες παρακολουθούν αυτά τα μέτρα που λαμβάνονται ή όχι σε εθνικό επίπεδο με τη δυνατότητα παρέμβαση και της ΕΚΤ. Θα ε, προσέθετα σε αυτά που σας είπα, είπα πως τα αντικυκλικά αποθεματικά που ενέκριναν οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι σε μηδενικά επίπεδα λόγω της κατάστασης ε, Δεν ξέρω ποιο γράμμα εννοείται, γιατί παίρνουμε πολλά. Μα εγώ προτείνω να το δημοσιεύσουμε. Θα, θα μας ενδιαφέρει, θα μας ενδιαφέρει όλους, πιστεύω, το περιεχόμενο, λέει ο κύριος Γκίγκολτ. Η κυρία Νουή, ναι, θα λέγανε και άλλα πολλά άμα τα δημοσιεύαμε. Τόσο πάνω τα περισσότερα είναι δημόσια όπως ή άλλωστε. Για το στρέφει για το δεύτερο πυλώνα, για να μην είμαστε προκυκλικοί, αφαιρέσαμε 25 μονάδες βάσης ε, για ε, όλες τις τράπεζες ε, στον SSM. The outcome of our exercise by 25 basis points uh, for every... Γιατί με μην ξεχνάτε ότι ε, χρειαζόντουσαν ηρωικά μέτρα και Δείτε και πω περιγραφει κατασταση στο εγγραφο της Ευρωπαϊκή επιτροπης οι τραπεζες ε, ξερουν πω εαν πλησιάσουν το, τα μέτρα του δεύτερου πυλώνα και μπουν στο, σε αυτό τον λόγο της έγκαιρης προειδοποίησης για τις απαιτήσει του δεύτερου πυλώνα με τις 25 μονάδες βάσης θα πάρουν γράμμα από εμά και θα τους προειδοποιήσουμε προσοχή προσοχή πλησιάζεται ε, το σημείο ενεργοποίησης και πρέπει να κάνετε κάτι για να αποκαταστήσετε την κατάσταση σε σχέση με τις κεφαλαιοχικές απαιτήσεις. Uh, Νομίζω ότι δεν έχουμε, ε, δεν έχετε αναλύσει το πλήρω το έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη δεν έχει αναλυθεί από την ενιαία υποπτική αρχή, αλλά αυτή είναι η κατεύθυνση που ακολουθεί. Πάντω αυτά δεν προέκυψαν από εκείνη την επιστολή των, από του λομπίστε. Μιλάμε για επαρκή επίπεδα κεφαλαιοποίησης ε, και θέλαμε να προσθέσουμε αυτή την άσκηση ε, 30 μονάδων βάσης. Ήταν λογικό και αυτό κάναμε. Για το λόγο που της ε, ε έγκαιρης προειδοποίησης, σημείο ενεργοποίησης έγκαιρης προειδοποίησης. Πρόεδρος, φυσικά είναι πολύ καλό να ακούμε τις εξηγήσεις από πλευράς τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατάλαβα εγώ σε ποιο γράμμα από λομπίστες αναφερόσασταν. Μάρκο Βάλι. Θα ήθελα, όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, να πω πως ε, είναι καλή αντίδραση αυτή να μην τρομοκρατηθούμε και να μην ε, ε, να, να αντιδράσουμε, να μην παραμείνουμε απαθείς. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις για την κυρία Νούη. Όπως είδαμε από την αρχή της κρίσης, τα ευρωπαϊκά όργανα προσπάθησαν να αξιολογήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ε, τα πιστοτικά ιδρύματα ε, στους κινδύνους στον τομέα των πιστοτικό και όχι των χρηματοδοτικό. Το σύστημα το τραπεζικό στην Ιταλία είναι θα έλεγα στραμμένο στην επιχειρηματικότητα και όχι σε άλλα τραπεζικά συστήματα ιδιαίτερα επικίνδυνα όπως στη Βόρεια Ευρώπη, στην Γερμανία όπου υπάρχουν ε, πολλές τράπεζες ε, με ε, υψηλά επίπεδα κινδύνου. Εμείς στην έκθεση για την Πιστοτική Ένωση που ψηφίσαμε στο Κοινοβούλιο κάνουμε διάφορες εκτιμήσεις σχετικά και με τη λειτουργία του SSM γιατί αν περιορίσουμε την προσοχή μας μόνο στους κινδύνους στον τομέα τον πιστοτικό τότε ίσως να διευρύνουμε την κακή εικόνα και σε πιο, με πιο σφαιρικό τρόπο. Θα ήθελα να μάθω λοιπόν αν υπάρχει επιθυμία από πλευρά σας ε, να λυθεί το πρόβλημα αυτό το χρηματοπιστωτικό, του κινδύνου του χρηματοπιστωτικού ή θέλετε μόνο να ασχοληθείτε με το θέμα το πιστωτικό και να αγνοήσετε τα συστημικά τελικά θέματα των τραπεζών, δηλαδή τα ενεργά τρίτου επίπεδου. Και τώρα σχετικά με το χαρακτηρισμό risk-free για τα κρατικά ομόλογα. Ε, είπατε ότι προτιμάτε να υπάρξει μια σταδιακή αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα λειτουργήσει αρνητικά για τις χώρες που έχουν υποστεί ιδιαίτερα αρνητικά στοιχεία στα πλαίσια της κρίσης που προηγήθηκε. Οπότε μήπως η αλλαγή του καθεστώτος αυτού να οδηγήσει σε μεγαλύτερα προβλήματα βάρη και κινδύνου στις χώρες οι οποίες έχουν ήδη χτυπηθεί και που δεν είναι και υπεύθυνε για την πιστοτική κρίση. Τώρα, στην Ιταλία υπάρχει το θέμα της συγχώνευσης των λεγόμενων και Popolari. Οι τράπεζες αυτές θα μπορούσαν με, θεωρητικά να οδηγήσουν σε μία, θα έλεγα, καλύτερη κατάσταση, από την άλλη όμως ε, τελικά αν ενώσεις δύο ευπαθείς και εύθραστες καταστάσεις αποκτά μια χειρότερη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρατήρησή σχετικά. Ε, μιλήσατε πιο πολύ για το πιστοτικό κίνδυνο. Κοιτάξτε, εστιάζουμε σε όλων των ιδίων τους κινδύνους για τις ε, τράπεζες και πράγματι κάνουμε αξιολόγηση της κεφαλαιοποίησης ε, των τραπεζών και προφανώς οι μικρότερες τράπεζες είχαν αυτούς τους ε, κινδύνους αλλά ίσως να μην φαίνονταν τόσο πολύ. Οπότε αν δει κανείς την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την αξιολόγηση των κινδύνων αυτών βλέπουμε πως είναι πάρα πολύ απαιτητική. Και πάλι λαμβάνουμε υπόψη κάθε είδους τραπεζικό κίνδυνο για να αξιολογήσουμε ε, τους μελλοντικού τραπεζικούς κινδύνους. Σημαντικό κομμάτι της δουλειά μας. Όσον αφορά τον κίνδυνο των κρατικών ομολόγων αναφέρατε την ανάγκη μιας αδιακής διαδικασίας και συμφωνώ πλήρω. Είναι δύσκολο ζήτημα. Θα χρειαστεί χρόνος, είναι κάτι το ευαίσθητο, το δύσκολο και ξεκινάμε με διαφορετική κατάσταση και αυτό ακριβώς κάνουμε ε, κάνουμε με την ισχύα μας. Η Επιτροπή της Βασιλείας ε, το κοιτάει και θα κάνει προτάσεις και μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δει πώς θα μεταφερθεί στο εθνικό δικαίωμα. Εσείς είστε οι νομοθέτες, όχι εγώ. Τα εργαλεία θα μου τα δώσετε εσείς. Δεν μπορώ να ξεκινήσω να αλλάζω τους ε, κανόνες του παιχνιδιού. Εγώ ακολουθώ τους κανονισμούς για την Ιταλική συγχώνευση που αναφέρατε. Πρόκειται για κάτι το πολύ σημαντικό και πρέπει να επιτύχει ακριβώς γιατί είναι η πρώτη μια σειρά ε, τέτοιων επιχειρήσεων. Και όλοι γνωρίζουμε σε άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη, ε, πως ε, και στην Ιταλία. Ε, διάφορες συγχωνεύσεις είχαμε που κατέληξαν ε, σε μεγαλύτερες δυσκολίες των τραπεζών που προέκυψαν. Οπότε συνεργαζόμαστε με τους ε, Ιταλούς συναδέλφους Ε, για να είναι ισχυρές οι τράπεζες και πρέπει να έχουμε μια κατάσταση συγκρίσιμη με, συγκρίσιμη με τις άλλες τράπεζες στην Ιταλία, όχι με άλλες χώρες. Και οπωσδήποτε καλωσορίζουμε και καλοδεχούμενες αυτέ οι συγχωνεύσει, αλλά πρέπει να είναι και επιτυχημένε. Και για να είναι επιτυχημένες υπάρχουν κάποιες απαιτήσει βεβαίω. Και εγώ θεωρώ πως αυτό έχει γίνει κατανοητό. Γιατί βλέπω στον τελικό τύπο ότι φέρομαι εγώ όσο το άτομο το οποίο φασίζει. Εγώ δεν έχω τέτοιε αρμοδιότητε. Υπήρχε ευρύτατη πλειοψηφία, πω και ομοφωνία όσον αφορά τις απαιτήσει που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Μπουρκχαρτ Μπάλτς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις. Κοιτάξτε τώρα η Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει το επιτόκιο αναφορά σε ένα ιστορικό χαμηλό. Είναι σε αρνητικά επίπεδα πλέον και εσείς ως επικεφαλής της ε, ΣΕΣΕΜ μιλήσατε για τον διαχωρισμό μεταξύ των λειτουργιών εποπτείας ε, και της ε, νομισματικής ε, πολιτικής. Μήπως έτσι λοιπόν μεταφέρουμε κάπου αλλού κινδύνους καθώς τα κλασικά επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών πλέον δεν είναι ανταγωνιστικά και θα πρέπει να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση του τραπεζικού κλάδου. Το δεύτερο ερώτημα η Ευρωπαϊκή Αρχή Διάσωσης ε, Τραπεζών ε, για το ΕΜΡΕ ορίζει ένα πανευρωπαϊκό στάνταρ τουλάχιστον 8% ε, και νομίζω πως συνεργάζεται στενά και θα έπρεπε να ακολουθείτε κοινή πορεία. Το ερώτημά μου είναι πώς θα στηρίξετε εδώ πέρα την συνάδελφό σας, την κυρία Κένιγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να σχολιάσω αυτό το επίπεδο, αφού είναι νομισματική πολιτική της έκτη. Αλλά όντω, αυτό που βλέπω είναι ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για την κερδοφορία των τραπεζών. Λόγω των ε, επιτοκίων. Είναι όμως και πλεονέκτημα για την ποιότητα του credit risk για ε, ε, κινδύνων της πίστης. Ε, θα μπορέσουν οι δανειστές λοιπόν, οι, δανειζόμενοι να, οι δικαιούχοι των δανείων να προστατευτούν καλύτερα. Ε, και μην ξεχνάμε ότι έχουν τα εργαλεία τους ε, οι τράπεζες κόστος προς εισόδημα παραδείγματο χάρη. Αν δούμε το λόγο το που παρουσιάζουν οι τράπεζες στην Ευρωζώνη παρατηρούμε διαφορές ιδιαίτερα υψηλό σε ορισμένε περιπτώσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχει περιθώριο για να έχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για να αντιμετωπίσουμε την πίεση επί τη κερδοφορία λόγω χαμηλών ε, επιτοκίων. Η ψηφιοποίηση επίσης Όλο ένα και περισσότεροι πελάτες, κυρίως της νέας γενιάς, ε, ζητούν ε, τις τραπεζικές υπηρεσίες ε, και ε, θα πρέπει να ακολουθήσουν ε, αυτή την κατεύθυνση για να μην απειληθούν από το FinTech. Αυτός ο λόγος λοιπόν του κόσμου προς το εισόδημα έχει ιδιαίτερη σημασία. Τώρα ο προσδιορισμός του ΕΜΡΕΛ από την ενιαία εποπτική αρχή, ναι, όντως πρέπει να συνεργαζόμαστε στενά με το ενιαίο Συμβούλιο Καθάρισης Τραπεζών. Πρέπει να τους δώσουμε τις απαιτούμενες προβολές για να κάνουν τη δουλειά τους. Εάν δεν είμαστε σίγουροι για το όριο ανάμεσα σε ότι πραγματικά χρειάζεται και τι όχι, ας είμαστε γενναιόδοροι. Καλύτερα περισσότερα να έχουν παρά λιγότερα και ειλικρινά. Η κυρία Κένικ ε, ήταν ιδρυτικό μέλος του SSM. Ε, γνωρίζει, κατέχει τη λειτουργία του, του μηχανισμού του ενιαίου μηχανισμού και πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι συζητούμε πολύ συχνά δυο τρει φορέ την εβδομάδα, θα έλεγα, κατά μέσο όρο. Μια χαρά λειτουργεί λοιπόν. Είναι ο πρώτος χρόνος πλούς λειτουργίας και είναι λεπτό το ζήτημα αυτό της δουλειάς του ενίου εποπτικού συμβουλίου. Σίγουρα, σίγουρα θα τους προσφέρουμε κάθε βοήθεια που μπορούμε. Ευχαριστούμε. Ο Μπερνάρ Μονό. Ε, Ευχαριστώ για την παρουσία σας, Πρόεδρε. Αυτή τη θλιβερή μέρα η πολιτική μου ομάδα και εγώ εκφράζουμε την συμπάθειά μας στα θύματα της τρομοκρατικής ενέργειας. Τώρα, στα πλαίσια της ε, νομοθεσίας ε, για την Τραπεζική Ένωση τίθεται το θέμα της διασφάλισης των πελατών και τι γίνεται σε σχέση με την πώληση του χρέους όταν προέρχεται αν κάτι τέτοιο εν πάση περιπτώσει θα διαμόρφωνε συνθήκες ε, οι οποίες θα επέτρεπε στους οικονομικούς εταίρους να κρίνονται με πανικό σε σχέση με τις αλλαγές της αγοράς. Λιγότερη πτυτικότητα λοιπόν και λιγότερος πανικός στις αγορές. Ξέρουμε ότι τον προηγούμενο μήνα υπήρξαν προβλήματα με τα ομόλογα κάποιων συστημικών τραπεζών που δεν θα πω το όνομά τους. τα προβλήματα με τις Ιταλικές τράπεζες το απέδειξαν μέχρι τέλους. Τα νοικοκυριά δυστυχώς έμειναν με τα χαριά στα χέρια μέχρι τη στιγμή ακριβώς που διαλύθηκαν οι τράπεζες αυτές με το άλοθη της προστασίας κάποιων κατηγοριών καταθετών στην ουσία επιβάλλονται κανόνες οι οποίοι οδηγούν στη μεταφορά των τοξικών τίτλων που θα χαθούν στην μεγάλη μαύρη τρύπα των δανειστών. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε το ναυάγιο αυτό. Μήπως αυτή το υποκείμενο χρέος θα πρέπει να αφορά μόνο τους θεσμικούς εμπλεκομένους και καταθέτες ή μήπως η τράπεζά σας θέλει να φροντίσει κυρίως τις ιδιωτικές τράπεζες και όχι τόσο τους καταθέτες και τους αποταμιευτές. Θα απαντήσω στα αγγλικά, λέει η κυρία στην ε, ερώτηση που έθεσε ο Γάλλος Ευρωβουλευτής. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία η ασφάλεια των ε, πελατών των τραπεζών. Τώρα αν το χρέος θα ε, πωλείται σε επίπεδο λιανικής ή όχι αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είμαι εγώ υπεύθυνη για τον καθορισμό αυτό. Οι υπεύθυνε αρχές για την εποπτεία της αγοράς στις 19 χώρες είναι αυτές οι οποίες αποφασίζουν τι μπορεί να απολυθεί σε επίπεδο λιανικής ή τι μπορεί να δοθεί σε επενδυτές, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με ομόλογα και άλλου είδους σύνθετα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή οι αποφάσεις αυτές έχουν ληφθεί για το αν θα απολυθούν σε επίπεδο λιανικό ή όχι. Υπάρχουν αρχές στις χώρες οι οποίες είναι υπεύθυνε για την προστασία των καταναλωτών και θα πρέπει οι αρχές αυτές να φροντίζουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν καταχρηστικές κινήσεις και να είναι υπεύθυνε για να εγκρίνουν το ποιος μπορεί να αγοράσει ή όχι τέτοιου είδους χρέος. Ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και έχω εμπειρία πάνω σε αυτό. Μετά το 2010 ήμουν υπεύθυνο και για τα θέματα αυτά στη Γαλλία αλλά στην παρούσα φάση αυτό δεν είναι τμήμα της ευθύνης την οποία έχω. Και δεν έχω καθόλου προσωπικό το οποίο θα μπορούσε να ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Δεν ανήκει στις αρμοδιότητες μου. Υπάρχει και η ΕΣΜΑ όπως ξέρετε, η οποία στην ουσία λειτουργεί πονδιακά για τις επιμέρους ε, ε, εποπτικές αρχές των τραπεζών των διαφόρων χωρών η Ένωση των Κεφαλαίων είναι κάτι το οποίο τελικά νομίζω θα ενισχύσει την προστασία των Ευρωπαίων επενδυτών. Τώρα μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εκδώσει συστάσεις. Όχι, αυτό δεν θα γίνει κατανοητό από την αγορά. Δεν θα πρέπει εμείς να, θεωρούμε, να θεωρηθούμε εισοδιστές σε τομείς οι οποίοι δεν ανήκουν στη δική μας αρμοδιότητα. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι οι επενδυτές θα πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένοι και δεν θα πρέπει να αγοράζουν πράγματα και προϊόντα τα οποία δεν κατανοούν. Νομίζω ότι αυτός είναι βασικός κανόνας. Αν δεν είναι κατανοητό το προϊόν δεν το αγοράζεις, είναι πάρα πολύ απλός ο κανόνας. Πέραν αυτού όμως εγώ όπως είπα δεν είμαι υπεύθυνη για αυτή την δύσκολη ευαίσθητη δραστηριότητα, αλλά είμαι πρόθυμη να βοηθήσω τους σεναδέλφους οι οποίοι έχουν τη συγκεκριμένη ευθύνη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε άλλωστε μία συνάντηση με τους συναδέλφους της ΕΣΜΑ και συζητήσαμε το θέμα αυτό. και του είπα ότι περιμένουμε πολλά από την ΕΣΜΑ έτσι ώστε οι επενδυτές να κατανοούν ότι μπαίνουν σε έναν δύσκολο κόσμο μετά την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας της EBRD σε σχέση επίσης και με τις δυνατότητες και πιθανότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν και ότι υπάρχει εγγύηση μέχρι τις 100.000 ευρώ. Πέραν αυτού όχι. Ευχαριστώ κύριος Φων Βάιστσακια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. less able to conduct a, a, a, a good and interesting hearing. Um, Madame uh, Nui, um... Κυρία Νουή, στην Επιτροπή μας ε, το 2016 συζητήσαμε βεβαίως ε, το... θα συζητήσουμε το θέμα της Ευρωπαϊκής εγγύησης, των Καταθέσεων και οπωσδήποτε θα συζητήσουμε και το σε ποιο βαθμό απαιτείται περαιτέρω μείωση των κινδύνων. Λοιπόν, έχω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Εάν θεωρείτε πως αυτό ισχύει όντως, τι θα έπρεπε δηλαδή να κάνουμε για να αποφευχθεί ένας πιθανός ηθικός κίνδυνος του έντις ε, και αν ισχύει αυτό τι, με, τι μορφή θα έπρεπε να έχουν αυτά τα μέτρα. Και ελπίζω να γίνει η συζήτηση να δούμε πόσο γενναιόδοροι θα είμαστε με την παροχή Έμπρελ. Υπάρχει η συζήτηση που ξεκίνησε ο Ντάισελμπλουμ για το θέμα του λόγου μόχλευσης. Τι θα κάνουμε με την έκθεση των κρατών. Βεβαίω είναι ένα συγκεκριμένο ερώτημα προς ε, σας το αγαπημένο μου θέμα, το θέμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων των τραπεζών και είδα ότι στο Baden Baden κάνατε μια παρουσίαση σε Γερμανούς επιχειρηματίες ε, για το θέμα αυτό και μάλιστα αναφερθήκατε στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τραπεζών ακριβώς για να αντιμετωπιστεί το θέμα της επιδότησης από τη Λιανική Τραπεζική των πιο επικίνδυνων δραστηριοτήτων. Και βέβαια μιλήσετε και για τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων αν αυτό είναι αναγκαίος. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το έντις την εγγύηση των ε, καταθέσεων Προφανώς ε, καλωσορίζουμε την ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης. Αυτό ακριβώς λείπει από την ε, Τραπεζική Ένωση και είναι θετικό το ότι γίνονται συζητήσεις. Είναι σημαντικό οι συνεισφορές των τραπεζών στο Ταμείο να βασίζονται στον κίνδυνο σε σύγκριση με όλες τις τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης, όχι μόνο στις τράπεζες της κάθε χώρας. Όσον αφορά τον διαμοιρασμό του κινδύνου, θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει αυτό παράλληλα με την οικοδόμηση του ΕΔΙΣ. Μια σταδιακή εισαγωγή του ΕΝΤΙΣ είναι αναγκαία για να λάβουμε υπόψη την διαφορετική αφετηρία του κάθε εθνικού συστήματος εγγύησης ε, καταθέσεων. Οπότε έτσι επιτρέπεται η σταδιακή εισαγωγή στο νέο σύστημα για να προχωρήσουμε σε έναν δίκαιο ανταγωνισμό στην Τραπεζική Ένωση και μείωση του κινδύνου. Θεωρούμε λοιπόν πως ε, η μείωση του κινδύνου και ο διαμοιρασμός του είναι στοιχεία που συμπληρώνονται και δεν θα πρέπει να είναι προαπαιτούμενα. Χρειάζεται τώρα ένα σαφής οδικός ε, χάρτης ε, για να πάμε σε ένα πλήρες εντύλ ε, στις φάσεις της ε, αντασφάλισης, ε, συνασφάλισης που βεβαίως είναι μεταβατικές φάσεις. Το τελευταίο κομμάτι, α ναι ναι, οι διαρθρωτικές ε, μεταρρυθμίσεις και τα πλέον εκτήματα του διαχωρισμού. Πριν από την κρίση υπήρχαν κάποιες ε, υπερβολές ε, στις δραστηριότητες της αγοράς του ε, είχαν αναλυφθεί. Οι τράπεζες που έκαναν αυτές τις λειτουργίες υπέφεραν κατά τη διάρκεια της κρίσης και μείωσαν σημαντικά οπωσδήποτε τις λειτουργίες τους αυτές. Αλλά μπορεί να υπάρχει πειρασμός ε, αν πιεστεί η κερδοφορία τους να επανέλθουν σε αυτές τις δραστηριότητες για να βγάλουν γρήγορα κέρδη αλλά βεβαίως αυτά εμπεριέχουν και έναν κίνδυνο ζημιών. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε αυτά τα ζητήματα. Τούτων λεχθέντων θεωρώ πως αυτά τα οποία έγιναν σε Γαλλία και Γερμανία π.χ. και σε άλλες χώρες ίσως είναι ένας καλός, ε, είναι ο σωστός τρόπος γιατί και πάλι ε, στην Ευρώπη μεταξύ λιανικής, τραπεζικής ε, και εμπορικών τραπεζών κτλ υπάρχουν αυτές οι λειτουργίες δημιουργίας αγοράς που θα μπορούσαν να πάνε σε μια ε, δραστηριότητα trading αλλά πάλι η χρηματοδότηση αυτής της δραστηριότητας θα είναι πιο ακριβή το κόστος για τους πελάτες θα είναι μεγαλύτερο θα υπάρχουν λιγότερες τέτοιες ε, δραστηριότητες ε. ή θα πάνε στις εμπορικές τράπεζες ως τμήμα των εμπορικών, της εμπορικής τραπεζικής εγώ έχω πολύ συγκεκριμένες απόψεις επί του θέματος. Τα όσα έγιναν είναι λογικά. Οι επόπτες έλαβαν ε, αρμοδιότητες για να αξιολογήσουν πότε υπάρχει ανάγκη διαχωρισμού και πότε όχι. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει άλλο ένα ερώτημα. Δεν ναι, ναι, έχουμε αργήσει όμως, λέει ο πρόεδρος. Υπερβάμος Μπερές. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητή Ντανιέλ Νουή. Γίνεται η πρώτη μεταρρύθμιση του συστήματος για τα λογιστικά πρότυπα και Όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο συνειδητοποιώ ότι καταρχάς είχαν κατά νου τους ε, τις τράπεζες ε, αυτοί που σκέφτηκαν την μεταρρύθμιση. Γιατί για τις ασφαλιστικές ε, θα έπρεπε να θέσουμε σε εφαρμογή αυτή την αρχή μέχρι ότου η ESB να φτιάξει και τα αντίστοιχα πρότυπα που θα ήταν προσαρμοσμένα στο τομέα των ασφαλιστικών εταιριών. Πέραν από αυτούς τους δύο γνωστούς τομείς. Έχουμε, παραδείγματος χάρη για τους ε, μακροπρόθεσμους επενδυτές, ε, ε, ανησυχίες για το EFRS ως προς την προκυκλικότητα των μέτρων και ως προς την ικανότητα αξιολόγησης των μακροχρόνων επενδύσεων κατά τον καταλληλότερο τρόπο. Εγώ το αντιλαμβάνομαι, ναι, έχετε, κοιτάζετε τα πράγματα από την τραπεζική οπτική γωνία, όμως ε, σίγουρα εξετάζετε και σφαιρικότερα την κατάσταση. Λοιπόν, δεν ε, συμφωνείτε ότι η νέα μεταρρύθμιση προσανατολιζόταν προς τις τράπεζες και ότι υπάρχουν και άλλες λογιστικές ανησυχίες ε, για την δίκαιη αξία για ολόκληρο το φάσμα των φορέων ε, της αγοράς που θα κληθούν να εφαρμόσουν τα νέα πρότυπα, όμως πρέπει να γίνει ένα προσαρμογή επάντηση, Δεν είμαι τόσο απεσιόδεξη για το IFRS 9. Ξέρω ότι πιστεύουν πολύ ότι αυτός ο λογιστικός υπολογισμός επί της ε, ε, δίκαιας τιμής θα επηρεαστεί με την εφαρμογή του νέου κανόνα του IFRS εμείς όμως δεν βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Για τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία έχουμε ε, το νέο μοντέλο για τις ζημιές ε, εφαρμόζοντας στο FRS 9 βασιζόμενοι στη διαφάνεια και στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Αυτές είναι οι νέες αρχές και το νέο μοντέλο εάν εφαρμοστεί σωστά κατά τη γνώμη μας, θα οδηγήσει πιο έγκαιρη προειδοποίηση των ζημιών αμβλύνοντας έτσι την ε, προκυκλικότητα του IES 39 ε, που ε, αντικαθίσταται πλέον. Για το νέο μοντέλο Edge Accounting ε, πιστεύουμε ότι θα μειωθεί η τεχνητή πτυτικότητα για τις απώλειες ε, μειώνοντας ε, την ψαλίδα των πολιτικών edging, βοηθώντας δηλαδή τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θετικό το FRS 9. Προς Μπορώ να σας πω ότι πολλές τράπεζες δεν ενθουσιάζονται για το IFRS 9 και λένε ακριβώς αυτό, ότι πρέπει να λάβουν περισσότερο υπόψη την παράμετρο της χρηματοοικονομικής σταθερότητας κατά την έγκαιρη τον έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση για τις εφαρμοστικές διατάξεις του IFRS 9 Θέλουμε να είναι ομαλή, εύρυθμη μετάβαση προς το νέο σύστημα. Δεν θέλουμε ξαφνικά να ανακαλύψουν οι τράπεζες ότι πρέπει να έχουν υψηλότερα αποθεματικά σε σχέση με αυτά που είχαν προβλέψει. Συνεργαζόμαστε μαζί του με του οικονομικούς ελεγκτές για να υπάρξει συνειδητοποίηση όλων των επιπτώσεων του νέου συστηματο. Εν γέννη πάντω, το εκλαμβάνουμε ως θετικό το νέο σύστημα και Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει αυτή τη νέα γραμμή, ούτως ώστε γέρος να μπορέσουμε ε, να περάσουμε στην ε, ταχύτερη δυνατή εφαρμογή. Σχόλια εκτός μικροφώνου της κυρίας Μπερές. Η κυρία Νοή λέει, όχι, δεν ε, καταλογίζω τίποτα σε κανέναν. αφού μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι πιστεύω. Ε, κάποια φορά μπορεί να πούνε οι τράπεζε άμα τι μα πιέζουν να προετοιμαστούμε για το IFRS 9 ενώ έχουμε χρόνο και δεν έχουν ληφθεί αποφάσει. Μόλις ληφθούν οι αποφάσει θα είναι ευκολότερο για μένα να φροντίσω ώστε να καταλάβουν οι τράπεζε ότι περνάει γρήγορα ο χρόνο και πρέπει να ετοιμαστούμε. μόνο. Ευχαριστώ κύριε Νοήτρη, σε ερωτήσεις σε σχέση με την δυνατότητα η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια θα έχει επιπτώσεις στους καταθέτες των τραπεζών σε τρία διαφορετικά θέματα, τρία διαφορετικά επίπεδα. Καταρχάς, μηδενικές ρήτρε στις υποθήκες από πλευράς ορισμένων πιστοτικών ιδρυμάτων έτσι ώστε να αποφύγουν να είναι αρνητικό το επιτόκιο υπάρχει η λεγόμενη ρήτρα μηδέν ή μηδενική ρήτρα. Ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό. Η ίδια ιδέα είναι η δυνατότητα ορισμένες χώρες ε, να χρεώνουν αρνητικά επιτόκια στους καταθέτες με τον ίδιο τρόπο που οι τράπεζες και αυτές υφίστανται για τις καταθέσεις τους στην κεντρική τράπεζα τα αρνητικά επιτόκια. Θα ήθελα λοιπόν και πάνω σε αυτό υπάρχουν αρκετές πολεμικές για την κάλυψη ε, των, ε, των οικονομικών δραστηριοτήτων ε, σε σχέση με τους πελάτες των τραπεζών. Θα ήθελα την άποψή σας γενικότερα για το προηγούμενο θέμα. Uh, πρώτα απ' όλα το Εποπτικό Συμβούλιο προσπαθεί να αντιληφθεί τα 19 συστήματα στεγαστικών δανείων σε κάθε χώρα. Ήδη αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ε, τις διαφορές επιτοκίων. Και βέβαια ε, το τελικό το ζήτημα είναι αν υπάρχει σωστή προστασία των καταναλωτών. Και βέβαια αυτό είναι στα χέρια των εθνικών αρχών, όχι της κεντρικής ε, τράπεζας. Για εμάς, ε, στην κεντρική τράπεζα, είναι πάλι ένα θέμα ρυθμιστικό. Δηλαδή, ποιο είναι το θέμα, πρόκειται για κίνδυνο πιστοτικό, κερδοφορίας, ποιο είναι το μέγεθος του κινδύνου, τι εποπτεία απαιτείται, για να κάνουμε σωστά την δουλειά μας ως εποπτική αρχή. Οπότε για την ώρα το μέγεθος ε, του κινδύνου δεν δικαιολογεί τίποτα άλλο από τη δικιά μας ε, την πλευρά. Οπότε και πάλι από μια εποπτική σκοπιά το θέμα είναι αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος συμπεριφοράς παραδείγματος χάρη αν ε, η προστασία των καταναλωτών δεν είναι επαρκής Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τελειώνουμε εδώ. Δεν υπάρχει χρόνος για και έτσι για τους προφανείς λόγους. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Λουί που ήρθε. Είχε αγγλικά. Σε μια στιγμή δύσκολη και έγινε η ακρόαση όπως προβλεπόταν η επόμενη. Θα γίνει στις 13 Ιουνίου. Πιθανότατα βεβαίω πριν από αυτό θα ζητήσουμε ε, να έρθετε σε κάποια συνεδρίαση και κλεισμένων των φύρων. Για την ώρα σας ευχαριστώ τη χρήσιμη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Και για τη δουλειά που κάνετε στο πρώτο έτος ε, των δραστηριοτήτων σας. Ευχαριστώ. va falloir camper au, il va falloir camper au Parlement alors.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 But it's your decision. Yeah. No, dear colleagues, uh, um, I think we gave a good sign uh, keeping our point in the agenda with Daniel Nui. Καλά κάναμε και διατηρήσαμε το το, σημείο στη μέση διατέξη με την Ντανιέλ Νουή. Τώρα ο, η Αντιπρόεδρος ε, αρμόδια για τους ε, τα θέματα ασφαλείας για προφανείς λόγους ε, είναι απασχολημένοι και ε, διάφοροι άλλοι που θα έπρεπε να συζητήσουν με την EBA ε, για αυτό το θέμα της εποπτείας δεν είναι διαθέσιμοι και οπότε προτείνω αναβολή του ζητήματος. Μέχρι να έρθει ολόκληρη η διαπραγματευτική ομάδα ζητούμε συγγνώμη. Αλλά Νομίζω ότι είναι η καταλληλότερη απόφαση. Λύεται τη συνεδρία. Δεν έχουμε άλλο σημείο, έτσι δεν είναι. Α. Η επόμενη συνεδρίαση Προς το παρόν ε, συνεδριάζουμε στις 3, αλλά θα έρθουν σε επαφή μαζί σας, θα δούμε τι θα αποφασίσουν, πώς θα συνεχίσουμε. Mr. Fox, yes. Fox, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξέρω ότι οι συναδέλφοι από την EBA έκαναν την προσπάθεια να έρθουν να μας μιλήσουν. Πόσοι βουλευτές είναι εδώ πέρα να τους περιμένουν. Εγώ γιατί ήρθα και καταλαβαίνω ότι πρέπει να αναβάλουμε το πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Δεν καταλαβαίνω γιατί αναβάλλετε τη συζήτηση. Μα έκανα τη διαβούλευση και ε, τα είπαμε τους συντονιστές και λάβαμε υπόψη κυρίως ότι οι συγκητές για αυτό το ζήτημα δεν είναι εδώ και είναι, πρόκειται για την επίσημη εξέταση από πλευρά του Κοινοβουλίου και πρέπει να συζητήσουν διαπραγματευτέ με την Επιτροπή. Η Επιτροπή δεν είναι εδώ για λόγου ασφαλείας. Α, ήρθατε εσεί. Φόξ δεν σχετίζεται δηλαδή με τις, τρομοκρατικέ τις επιθέσεις. Ε, δεν είναι εδώ οι συγητές. Μα συνδέεται, ε, δεν είναι εδώ οι συγητές ε, για λόγους που συνδέονται με τις έκτακτες περιστάσεις που ζούμε όλοι τώρα. Κυρίως ο κύριος Σταγιάννη δεν Τέλο πάντων, βλέπετε τώρα, κοιτάξτε γύρω σας, δεν ε, είναι εδώ πέρα τα μέλη που έπρεπε να μιλήσουν. Οπότε κρίνω ότι είναι προσφορότερο να αναβάλουμε τη συζήτηση αυτού του ζητήματος. Και αυτή την απόφαση έλαβα.